επανεκμή επανεκβιομηχάνησης υπό το φω των πρόσφατων υποθέσεων Κατερπιλάρ και Άλστομ. Παρευρίσκονται το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον Υπουργό κύριο Κόρτσοκ και σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχετε το λόγο Υπουργέ. I So once again, Madam uh, President, uh, honorable members, Κυρία και κύριοι, αξιότιμα μέλη, κυρία Επίτροπε. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, διότι δεν θα παραμείνω καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης δυστυχώς, διότι πρέπει να επιστρέψω επιγόντως. Ολοκληρώνουμε τις διαπραγματεύσεις για τη Σύνοδο Κορυφή στην Βρατισλάβα. Τη Δευτέρα προσθέσατε στην ημερήσια διαταξή του το, το θέμα, γι' αυτό άλλαξα το πρόγραμμά μου γιατί ήταν σημαντικό να παρουσιάσω τη δήλωση. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραμείνω καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Τα νέα ε, που έφτασαν πολύ πρόσφατα στο Βέλγιο και την ε, Γαλλία για εργοστάσια που κλείνουν, δημιούργησαν, προκάλεσαν φόβο και αγωνία στις περιοχές. Οι πρόσφατες περιπτώσεις Κατεπυρά και άστρομ είναι ε, αντανάκλαση ενός ε, γενικότερου φαινομένου μαζικών απολύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αλλάζει το οικονομικό περιβάλλον με βαθιές επιπτώσεις στην ανεργία και κοινωνικές. Και στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη χαλιβουργία είχαμε πρόσφατες εξελίξεις και στη ΣΕΛ πρόκειται να υπάρξει μεγάλη αναδιάρθρωση άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να το κοιτάξουν αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να αφήσουμε να μας ξεφύγει αλλού η τεχνογνωσία μας και η βιομηχανική ή να αναλάβουμε αποφασιστική δράση για να βελτιώσουμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι βιομηχανίες μας. Τον Ιούνιο του 2013 Ήδη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αναγνωριστεί η ζωτική σημασία να υπάρχει μια ισχυρή οικονομική και βιομηχανική βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ε, στο ψήφισμά σας του 2014 τονίσατε ότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα αναφερθώ σε αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζητούν μια φιλόδοξη και ενεργή ε, βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να ε, υπάρχουν και κλαδικές πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανταγωνιστικότητα και για διατήρηση βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα θα πρέπει η ανταγωνιστικότητα αυτή η βιομηχανική να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις σχετικές πολιτικές. Υποδομές και ψηφιακές χρειάζεται να αναπτύσσονται και με μακροπρόθεσμη προοπτική. Η αγορά εργασίας επίσης να προβλέπει την ανάπτυξη και την απασχόληση και να καλύπτει και τα κοινωνικά δικαιώματα. Στη χρηματοδότηση έχει δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ε, που βοηθάει. Παρ' όλα αυτά ε, θα πρέπει να αρθούν και άλλα εμπόδια που παραμένουν έτσι ε, ε, να υπάρχει μια χρηματοδότηση από άλλες πηγές και ιδιωτικές και με δανειοδότηση. Υπάρχει Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων που συνεισφέρει και εκείνη. Τα δύο τρίτα των επενδύσεων αφορούν αποφάσεις που λαμβάνονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να συνεννοούνται με τη βιομηχανία. Οι περιφέρειες μπορούν να παίξουν εδώ ρόλο κλειδί για τον εξυγχρονισμό. Μεταξύ άλλων, αυτό μπορεί να γίνει με ε, την περιφερειακή πολιτική και τη βιομηχανική πολιτική να συνδέονται μεταξύ τους. Όπως έδειξαν οι πρόσφατες εξελίξεις, χρειάζεται και αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος, όπου να συμμετέχουν και κυβερνήσεις και κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ένωσης ε, αυτό ε, είναι πλέον γεγονός και το έχουμε κατανοήσει. Θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα κοινωνικοί εταίροι. Καλωσορίζει το Συμβούλιο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα που τους αφορούν άμεσα. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κάποια οικονομικά στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει έργα για την απασχολησιμότητα και έτσι ώστε να καταπραϊνθούν κάπως οι κοινωνικές επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων και να ανασυγκροτήσεων. Υπάρχει και το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης που απορροφά κάποιους κραδασμούς. Είναι όμως ένα εργαλείο ε, για να απαντά εκ των υστέρων σε τέτοιες καταστάσεις. Θα πρέπει από κοινού να ε, καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το σωστό πλαίσιο, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και διατηρώντας πάντα ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Κυρίε και κύριοι, η έρευνα, η καινομία, η ε, αριστεία είναι βασικά συστατικά της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούν εκπροσώπους ε, της ερευνητικής κοινότητας, της καινοτομίας και των επιχειρήσεων σε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη για την επανεκβιομηχάνηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πρατισλάβα στις 26 με 28 Οκτωβρίου και θα επικεντρωθούμε στην ανατεχνολογία, ε, στα προηγμένα υλικά, σε τεχνολογίες παραγωγής, κατασκευών και βιοτεχνολογία. Ένα άλλο στοιχείο κλειδί είναι η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας που έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Δυστυχώς ακόμα ε, δεν είναι συνεχτική η ανάπτυξη σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη, περιφέρειες, Ευρωπαϊκή Ένωση και η βιομηχανία έχουν να παίξουν όλοι το ρόλο τους στην ψηφιοποίηση και στην ανάπτυξη της βιομηχανικής διάστασης της ψηφιακής ε, ατζέντας θεματολογίου. Γι' αυτό υπάρχει και αντίστοιχη ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο, όπω έχει δηλώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο θεματολόγιο για τι νέε δεξιότητε, χρειάζεται πάντα εκπαίδευση, κατάρτιση και καλύτερη προσαρμογή των προσόντων και των δεξιοτήτων στι ανάγκε τη αγορά. Έτσι ώστε να υπάρχει ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και εργασία. Αξιότιμοι βουλευτέ, ε, είναι πολυσχηδή αυτή η προσπάθεια θέλουμε να επανεκβιομηχανίσουμε την Ευρώπη. Και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν εργάζονται σκληρά προς το σκοπό αυτό, αλλά και το Συμβούλιο. Η επανεκβιομηχάνηση θα απασχολήσει στις 29 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας και σας θυμίζω πάλι τη διάσκεψη του Οκτωβρίου στην Πρατισλάβα και σας καλώ να παρευρεθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που θα χρειαστεί να αποχωρήσω, αλλά ήδη έχω καθυστερήσει πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Βεβαίως το προσθέσαμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη κάπως καθυστερημένα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Τάισεν από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Οι πρόσφατες δηλώσεις από την Alstom και την Caterpillar για το κλείσιμο μεγάλων σημαντικών εργοστασίων στην Ευρώπη έχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, για τους ε, εργαζόμενους αλλά και για όλη την περιοχή στην οποία βρίσκονται. Είναι πολύ σημαντικό το ότι εδώ οργανώνεται αυτή η συζήτηση ιδιαίτερα σε σχέση με το μέλλον της εκβιομηχανίας και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να στηρίξουμε αυτούς που πλήττονται άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν προοπτικές προσανατολισμοί για τους εργαζόμενους οικογένειές τους, αλλά και για την οικονομία των περιεχών που πλήττονται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε όλα τα επίπεδα να στηρίξουμε αυτούς τους εργαζόμενους που έχασαν τις δουλειές τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτήν την πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν. Έχουμε σήμερα ηθική υποχρέωση να βρούμε λύσεις για αυτές τις περιοχές και αυτούς τους οικονομικούς κλάδους οι οποίοι γνωρίζουν αυτές τις αναδιαρθρώσεις. Είναι σαφές ότι καμία επιχείρηση δεν πρέπει να αποφύγει τις ευθύνες της έναντι των εργαζομένων. Διότι οι απολύσεις, το κλείσιμο ενός ε, εργοστασίου σαφώς και θα πρέπει να ακολουθείται από την αλληλεγγύη, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και την οικονομική στήριξη που διατίθεται για τους εργαζόμενους σε αυτές τις ε, περιοχές που πλήττονται. Και αυτό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και από την ε, επιχείρηση Caterpillar και από άλλες περιοχές στην περιοχή και επιπλέον στήριξη από το Ταμείο αυτό το Ευρωπαϊκό για την αντιμετώπιση της, ε, των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, αλλά υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης ε, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν στήριξη, σαν κατάρτιση για τους εργαζομένους, το ίδιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής, που θα πρέπει να συνδράμουν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Από την άλλη θα πρέπει να δημιουργηθεί και μία task force, μία ομάδα εργασίας από κοινού με τις αρχές του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να στηρίξουν όλους αυτούς ε, οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια δίνοντάς τους νομικές συμβουλές. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε έτσι ώστε αυτό που από την αρχή έχει στείλει σαν μήνυμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή την ανάγκη να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη, της ε, οικονομίας στην Ευρώπη, να υλοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2016. 20,4 δις διατίθενται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για επενδύσεις σε τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία και 150 δις 115 δις, συγγνώμη, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί στην ε, ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ, θα διατεθούν για να διπλασιαστεί το συνολικό ποσό που θα διατεθεί σε επενδύσεις ε, μέχρι το 2020 στην Ευρώπη. Σκοπός μας είναι να ακυρώσουμε τις δυσκολίες, να βγάλουμε όλα τα εμπόδια στην πρόθεση όλων αυτών των κονδυλίων στην πραγματική οικονομία, να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει όλη την επενδυτική και οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό στις προσπάθειές μας να διευκολύνουμε με καλύτερη ρύθμιση την λειτουργία των χρηματαγορών του τραπεζικού συστήματος, αλλά δημιουργώντας μέσω της νέας ατζέντα της Ευρώπης για νέα προσόντα νέες δυνατότητες κατάρτισης. Οι νέες δεξιότητες είναι κάτι το οποίο σαφώς και θα ενισχύσουν την ε, ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την ευρωπαϊκή καινοτομία. Με αυτές τις επενδύσεις θέλουμε να βγούμε από τον φαύλο κύκλο της ανεργίας, δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης. Και αυτό προς τους νέους, προς τους ηλικιωμένους, προς τους άνεργους και προς όλους αυτούς οι οποίοι αλλάζουν θέσεις εργασίας και τομείς. Ο Τομέα ο βιομηχανικό στην Ευρώπη είναι ισχυρό. θα πρέπει όμω παρόλα αυτά να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσει, οι οποίε διαρκώ ε, εμφανίζονται και να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη παραμένει ανταγωνιστική, ελκυστική για την βιομηχανία. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κυρία Πίτροπη. Αρχίζει τώρα η συζήτηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Κυρία Γκροστάτ, πρώτα ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, δυστυχώς για άλλη μια φορά ξανασυζητάμε για αυτή την βαθιά κρίση έλλειψη επενδύσεων και ανταγωνισμού για την βιομηχανία μας στην Ευρώπη. Το κλείσιμο της Κατρεπίλα και της Άστρομ δείχνουν ακριβώς την κακή βιομηχανική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Έχουμε περισσότερα κλεισίματα από δημιουργία νέων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι ενσυχητικό και προκαλεί στον κόσμο θυμό και αγωνία. Παρ' όλα αυτά γνώριζε το κοινό την δύσκολη κατάσταση αυτών των επιχειρήσεων. Δυστυχώς όμως αναστήθηκε εσπευμένα και βιαστικά ένα σχέδιο σωτηρίας. Χωρίς να κοιτάξουμε ένα γενικότερο πλαίσιο πρόθεση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μας και δημιουργίας ενός κατάλληλου πλαισίου. Στην ουσία, οι επιχειρήσεις χρειάζονται αναδιάρθρωση για να προσαρμοστούν στις αλλαγές και για να αναπτυχθούν χρειάζονται ένα περιβάλλον κοινωνικό και φλοικό ευνοϊκό και να μην παραλύονται από τους μεν και τους δε. Στην περίπτωση της Alstom που γνωρίζω μου φαίνεται επικίνδυνο μια κυβέρνηση να προτείνει σε άλλη γαλλική επιχείρηση που αντιμετωπίζει δυσκολίες και έχει χρέη, την SNCF, προτείνει λοιπόν να κάνουν παραγγελίες βιαστικά, τεχνητές ψεύτικες παραγγελίες, ενώ εδώ και πολλά χρόνια στην Γαλλία δεν υπάρχει συνδρομική πολιτική. Αυτό λοιπόν που λείπει στην Ευρώπη είναι η πρόληψη. Μιλάμε συνεχώς για βιομηχανική πολιτική. Ποιος όμως προτείνει πραγματικές στρατηγικές βιομηχανικής ανάπτυξης μακρόπνοης για τις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις. Αυτό λείπει λοιπόν και δυστυχώς υποφέρουν οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν να κάνουν πολλά μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και στο κοινωνικό ντάπινγκ που υπάρχει στην Ευρώπη. Το κλείσμα αυτών των επιχειρήσεων λοιπόν αποτελεί κάτι το δύσκολο για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό είναι σημαντικό, όπως είπατε Επίτροπε, είναι σημαντικό να προστατευτούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Η βιομηχανία μας, αυτό που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Σταθερότητα φορολογική, σταθερότητα νομοθετική χρειάζεται να ενθαρρυνθεί από μακρόπνοες στρατηγικές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκροστέτ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Αγενά, για ένα μισή λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κλείνει λοιπόν, όπως ανακοίνωσε η κατέπειρα στον Κοσλή, πάνω από 6.000 εργάτες βυθίστηκαν στην έλλειψη κατανόησης και στην απόγνωση. Δεν είναι μοναδική περίπτωση. Φιλανδία, Nokia, Microsoft, πάνω από 8.000 απολύσεις. Σουηδία, Ericsson, πάνω από 1.500 απολύσεις. Κάθε εβδομάδα ε, υπάρχει ένα αίτημα για ενίσχυση από το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης. Το θέμα δεν είναι ότι κλείνει μια επιχείρηση, αλλά πώς κλείνει και γιατί. Η Καταλπιρλάρ είναι ένας όμιλος που ε, πηγαίνει και που πληρώνει λιγότερο. Στην Ελβετία πάει για να μην πληρώνει φόρους στην Ευρώπη. Επίσης είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση που επιλέγει να ανταμείψει το κεφάλαιό της παρά να επενδύσει σε στρατηγικές που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Είναι επίσης ε, κέντρο λήψης αποφάσεων εκτός της Ευρώπης ε, που παραγνωρίζει και αγνοεί ουσιαστικά τους εργαζομένους και τις υποχρεώσεις που έχει. Αυτό το βλέπουμε σε πολλές πολυεθνικές σήμερα. Η Caterpillar επίσης έχει και άμεση, είναι και μια άμεση επίπτωση της λιτότητας γιατί έχουν μειωθεί τα δημόσια έργα και υπάρχουν και λιγότερες επενδύσεις σε μηχανήματα. Ε, και πού είναι η πράσινη ανάπτυξη, ε, τι να κάνουμε τώρα. Κυρία Επίτροπε, το είπατε και εσείς, πρέπει να βοηθήσουμε τους εργαζομένους, τους απολυμμένους και τις ε, περιφέρειες που πλήττονται και ξέρω σε ποιο βαθμό εσείς είστε πρόθυμοι να το κάνετε. Δεύτερον, αναζωγόνηση των δημοσίων επενδύσεων και τρίτον, εκεί ε, που παράγεται ο πλούτος να ε, φορολογείται η επιχείρηση και να μην έχουν ε, απόλυτη ασυδοσία οι ξένοι επενδυτές. Εδώ είμαστε πρόθυμοι στο Κοινοβούλιο να δεχτούμε ιδιωτικά διατητικά δικαστήρια που θα αφήνουν να αλωνίζουν με ασυδοσία οι ξένοι επενδυτές. Και τέλος θα πρέπει να γίνουν μελέτες αντικτύπου για την παγκοσμιοποίηση και όχι μόνο για τα θετικά το ξέρω ότι υπάρχουν και θετικά. Είναι γεγονό. Αλλά και για τα αρνητικά. Το να αρνούμαστε ότι υπάρχουν αρνητικέ συνέπειε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε για να προσαρμοστούν και οι επιχειρήσει και οι δομέ μα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο ειλικρινεί ω προ την παγκοσμιοποίηση. Σα ευχαριστώ. Και εγώ. Η κυρία Στέβεν έχει το λόγο. Για μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρώτη σκέψη όταν ακούς μια τέτοια ανακοίνωση τύπου κατελπίλα ε, είναι για ε, τους απολυμένους. Ε, το κόμμα μου, NVA και η ομάδα μου, ECR, συμπάσχουν με τους απολιμένους εργαζομένους, διότι εκείνοι θα πληγούν περισσότερο από την κρίση αυτή. Ανησυχούμε πολύ για την παγκοσμιοποίηση. Η σωστή απάντηση είναι πολιτική, στοχευμένη και όρημη. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι κρίσιμα δεν θα πρέπει να υποκύψουμε σε προστατευτικές τάσεις. Η διεθνής ε, ανταγωνιστικότητα και ανταγωνισμός τελικά οδηγεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας, όχι λιγότερες. Θα πρέπει η ασφάλεια της εργασίας να προέχει σε σχέση με την ασφάλεια των θέσεων εργασίας. Ε, χρειάζεται προσαρμογή στην αγορά εργασίας με τη νέα τεχνολογία για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ευημερία μας, την εργασία μας και να τη βελτιώσουμε. Κανένας δεν περισσεύει στην αγορά εργασίας, ούτε είναι εξοφλημένο για λόγου ηλικία. Επειδή γυράσει και ο πληθυσμό, θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και απασχολούμε του πιο μεγάλου εργαζομένου. Πολλοί περιμένουν ε, από το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση στήριξη για τι ομαδικέ απολύσει. Αλλά το θέμα δεν είναι να πάει ο λογαριασμό στο φορολογούμενο. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας με μεταφορές πιστώσεων από τη μια χώρα στην άλλη. Χρειάζονται διαρθωτικές μεταφο... Ε, μεταρρυθμίσεις από τις χώρες και η χώρα μου σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό η κυβέρνηση δίνει το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Thank you. Madam Stevens, Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ταραμπέλα, μπλε κάρτα. Τι δέχεστε. Ο κύριος Ταραμπέλα. Άκουσα κυρία Στέβενς ότι είστε αλληλέγγυοι προς τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να δείξει κανείς την αλληλεγγύη του είναι όπως το κάναμε πριν από λίγα χρόνια στο Βέλγιο. Με εθνική αλληλεγγύη προτείναμε σε όλους να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα. Η ΕΛΒΑ σήμερα δεν βλέπω να προτείνει κάτι τέτοιο. Ίσως θα ήταν μια λύση. Γιατί είστε αντίθετοι προς την ε, πρόορη αυτή συνταξιοδότηση για τους εργαζόμενους αυτούς. Αγαπητέ συνάδελφε, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, αλλά να ακούτε αυτά που λέω κιόλας. Είμαστε κατά ε, του αποκλεισμού των ε, πιο ηλικιωμένων εργαζομένων. Εμείς είμαστε κατά της προσύνταξης, γιατί δεν είναι λύση. Θα πρέπει και οι πιο μεγάλοι εργαζόμενοι να μετεκπαιδεύονται για να μπορούν να βρίσκουν νέα δουλειά και όχι να βγαίνουν προώρα στη σύνταξη. Αυτό θέλουμε εμείς. Η προώρη συνταξιοδότηση δεν είναι σε καμία περίπτωση λύση. Αυτό είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεπρέ έχει το λόγο. Για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επίτρεπε, τις στι 2 Σεπτεμβρίου η Caterpillar ανακοίνωσε το κλείσιμο του εργοστασίου Τσοκοσία. Αυτό έγινε πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι καθώς και οι πολιτικοί βρίσκονται σήμερα μπροστά σε αυτήν την απόφαση και νομίζω ότι πλήττονται συγκεκριμένα χιλιάδες άνθρωποι άμεσα και έμεσα υπεργολάβοι και εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Το θέμα αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ε, απάνθρωπου καπιταλισμού. Βλέπουμε ότι η δίκηση της ε, επιχείρησης δεν απαντά είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική. Τους καλέσαμε και στο, στο Βελγικό Κοινοβούλιο, χωρίς όμως ανταπόκριση. Η κατάσταση είναι τραγική για μια περιοχή με πάρα πολύ υψηλή ανεργία, και με πολύ λίγες δυνατότητες ε, για απασχόληση. Βλέπουμε σήμερα ότι αυτό το σύμφωνο σταθερότητας έχει δέσει τα χέρια των κυβερνήσεων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Η Caterpillar σήμερα καλείται να ακολουθήσει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Ρενό. να δικαιολογήσει την απόφασή της για το κλείσιμο ενός εργοστασίου το οποίο είναι κερδοφόρο σε μια επιχείρηση που έχει θετικά αποτελέσματα. Δεύτερον, θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές που να προσφέρουν τα συνοδευτικά μέτρα και τις αποζημιώσεις που πρέπει στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα όλοι οι συνδικαλισ... όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν κινητοποιηθεί. Θα πρέπει και εμείς να στηρίξουμε τις προσπάθειες των εργαζομένων να μπορέσουν να απορροφηθούν από κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Όμως όλα αυτά δεν φτάνουν. Άκουσα σήμερα το πρωί τον πρόεδρο της Επιτροπής στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης που αναφ φέρθηκε σε μια Ευρώπη που προστατεύει, σε μια κοινωνική Ευρώπη. Θα ήθελα πολύ όλοι οι εργαζόμενοι της Κατερπίλαρ να νιώσουν ότι τους προστατεύει η δική μας Ευρώπη και ότι σήμερα τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι καθαρά αντιλαϊκά και αντικοινωνικά. Κυρία Πρόεδρε, ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να είναι συστατικό της Ευρώπης. Θα πρέπει να βρούμε νέα μέσα, νέα εργαλεία, όπως ένα ταμείο στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα το βιομηχανικό, που να στοχεύει τη βιομηχανία και οι επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στις χώρες μας να έχουν ένα κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς πιο δεσμευτικό και να τους περιορίζει τέτοιου είδους αποφάσεις για κλεισίματα εργοστασίων. Το σχέδιο Juncker με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει πραγματικά να είναι παραγωγικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέντελ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτρεπε, κυρίε και κύριοι, Επιτροπή θέτει φιλόδοξους στόχους για επαναβιομηχανοποίηση της ε, Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά εδώ βλέπουμε όχι μόνο την Caterpillar, αλλά και άλλες επιχειρήσεις που καταστρέφουν θέσεις ε, απασχόλησης, δυστυχώς. Και πολλές φορές βλέπουμε επιχειρήσεις οι οποίες ε, παίρνουν τέτοιες αποφάσεις ενώ είναι κερδοφόρες. Βεβαίως, στις περισσότερες ε, περιπτώσεις αυτές οι καταστροφές θέσεων απασχόλησης συμβαίνουν σε κερδοφόρες επιχειρήσεις. Αν κοιτάξει κανείς λίγο πιο μακροπρόθεσμα και αν κοιτάξει τους βιομηχανικούς τόσους σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στον τομέα που μας απασχολεί σήμερα, αλλά και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Και σήμερα βλέπουμε ότι η Alstom δεν είναι εξαιρέσει και στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Εδώ βλέπουμε ότι μειώνονται οι θέσεις απασχόλησης και σήμερα χρησιμοποιούνται τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Ταμείων, όπως το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, για να στηρίξουν τέτοιες κερδοφόρες επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν αποφάσεις περιορισμού των θέσεων αποσχόλησης. Θα σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμπερτς. Συνάδελφοι πιλέρ, μεταξύ 2009 και 2015 είχε πάνω από 5% αύξηση των μερισμάτων και 15% απόλυτη θέσεων εργασία. Αυτές οι Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς ότι ο καρκίνος της ε, παγκοσμιοποίησης ε, διαβρώνει την οικονομία μας και αντί για την ε, μεγέθυνση το κέρδος παραμένει το α και το μέγα των πολιτικών και βεβαίως δεν υπάρχει καθόλου ανταπόκριση στις κοινωνικές προσδοκίες. Είχαμε από το 2000 από το 20% μείωση στο 15% του πληθυσμού. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να προωθήσει τις ε, εμπορικές συμφωνίες, όμως θα πρέπει επίσης η Κομισιόν να ζητήσει βεβαίως και προσαρμογή στο Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν έθεσαν το στόχο της αύξησης του μεριδίου της μηχανίας στο ΑΕΠ είναι σωστό αυτό, γιατί είτε έχουμε να κάνουμε την ενέργεια, με την κινητικότητα, με τι οικοδομέ, η βιομηχανία έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά τη μετάβαση τη οικονομία μα προ μια οικονομία με χαμηλή χρήση πόρων και ενέργεια. Οπότε λοιπόν έχουμε κάθε συμφέρον ως εμείς και η Κομισιόν να καθοδηγήσουμε αυτή τη μετάβαση. Πέρα λοιπόν από τα συναισθήματα που προκαλεί το κλείσμα αυτών των επιχειρήσεων, θα πρέπει να μάθουμε αυτό το δίδυγμα και να δούμε ακριβώ τι γίνεται με τι πολιτικέ, τι βιομηχανικέ. Θα πρέπει καταρχά να δούμε τι θα κάνουμε με τα χρηματοοικονομικά. Έχουν πολλά, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Όσο το κέρδο ε, καθορίζεται από επιχειρήσει, οι οποίε είναι πολύ μεγάλε για να α, πέσουν, ε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Μετά θα δούμε την εμπορική πολιτική. Θα πρέπει να σταματήσουμε τα σχέδια εμπορικών συμφωνιών που εξυπηρετούν μόνο τους μετόχους και θα πρέπει να υποβάλουμε την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά σε όρους και προϋποθέσεις κοινωνικές και περιβαλλοντικέ. Μετά, η βιομηχανία θα πρέπει βέβαια να υπηρετεί την μετάβαση και η μετάβαση ακριβώ και την ίδια τη μηχανία. Έχουμε μέσα για να βάλουμε τη μηχανία μα ακριβώ στην, ε, μπροστά στην πρωτοπορία. Να έχουμε λοιπόν, όμω τα μέσα στη διάθεσή μα για να το κάνουμε αυτό. Το σχέδιο επένδυση Juncker αντί να μοιράζει από εδώ και από εκεί τα χρήματα, θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βιομηχανία και στην οικολογική μετάβαση. Και τέλος, τέλος, η βιομηχανία μας όλο και περισσότερο η βιομηχανική απασχόληση υποκαθίσταται από μηχανήματα. Δεν απαραίτητα κακό, υπό τον όρο ότι τα κέρδη βεβαίω θα πρέπει να κατανείμονται μεταξύ όλων. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ε, εργασία, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την κατανομή ε, εργασία και ε, κερδών. Διαφορετικά θα έχουμε μεγάλε απώλειε όσον αφορά τι θέσει εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λάμπερτ, ο κύριο Σαφχάουζερ θα ήθελα να σα κάνει μια ερώτηση. Με τη διαδικασία τη μπλε κάρτα, δέχεστε την ερώτηση. Κύριε Σαφχάουζερ, κύριε Λαμπέρτ, σα άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον πριν εκλεγώ εδώ βουλευτής, με κάποιους άλλους προέδρους των μεγάλων δημοσίων τραπεζών ζητούσαμε ένα σχέδιο επενδύσεων χρησιμοποιώντας τις διευκολύνσεις κεντρικής τράπεζας. Δισεκατομμύρια ε, που επενδύονται στις βιώσιμες ε, οικονομίες και την πράσινη οικονομία. Γιατί δεν υιοθετείτε αυτή την ιδέα. Μήπως χρειάζεται ευρωπαϊκός προστατευτισμός τουλάχιστον για να υπάρχει μια στοιχειώδης αμοιβαιότητα ε, στο άνοιγμα των αγορών. Κοιτάξτε, έχω δυόμιση λεπτά, αγαπητέ συνάδελφοι. Δεν λέω όλε τι ιδέε, γιατί δεν μπορώ να τα πω όλα, δεν τα προλαβαίνω η μαζική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ποσοτική χαλάρωση, διαρκεί χρόνια και καταρκεματίζεται με τρόπο τελείως αδιάκριτο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό εμείς ζητούμε να υπάρξει ένα πρασίνισμα, δηλαδή είναι στοχευμένες οι επενδύσεις. Βλέπουμε ότι εκρήγνεται αγορέ αγορές ε, ρευστών γιατί υπάρχουν ενέσει ρευστότητα, αλλά λέμε να εστιάσει εκεί και αυτή η τράπεζα και άλλε δημόσιε τράπεζε επενδύσεων η ρευστότητα αυτή να πάει στην πράσινη οικονομία και στη μετάβαση εκεί. Είναι προφανές και αυτονόητο, παρόλα αυτά ε, ε, λείπει ακόμα η πολιτική βούληση. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε πλειοψηφία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να υλοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικολάς Μπέ έχει το λόγο. Η υπόθεση του εργοστασίου Alstom στον Πελφόρ που ελπίζουμε ακόμα να είναι πιο ευνοϊκή στην έκβαση από ό,τι τα χαλιβουργία στον Καντράνς και στο Φλωράνς είναι εμβληματική για την υποταγή των ηγετών μας στις επιταγές των ε, μετόχων και των ε, συνταξιδοτικών ταμείων. Ο οποίος συμβολισμός για το εργοστάσιο αυτό άνοιξε το 1879 και το 1971 βγήκε το πρώτο πρωτότυπο του τρένου υψηλής ταχύτητάς μας το ε, ε, περίφημο ΤΖΒ, για το οποίο όλος ο κόσμος μαζιλεύει, μέχρι 9.000 εργαζομένους. Σήμερα στον τριτογενή τομέα δεν γίνονται προσλήψεις, ενώ καταστρέφονται στη βιομηχανία. 33.000 πέρσι μόνο στη Γαλλία. Δεν είναι άμυροι ευθυνών οι ηγέτες μα, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιβάλλει τη μετάβαση της οικονομίας μας στη χρηματοοικονομία. Και υποτίθεται ότι είναι ε, ελεύθερος ο ανταγωνισμός και εν ονόματι αυτού μας Αγορεύει κάθε ε, προστατευτισμό, ακόμα και ευρωπαϊκό. Και υποτίθεται ότι για να μην υπάρχουν ε, μονοπόλια πρέπει να διαχωρίσουμε στο σιδηρόδρομο το δίκτυο από τη λειτουργία του. Έτσι λοιπόν σαλαμοποιούν τις εταιρείε μας για να τις πουλήσουν και έρχεται εδώ να συνεχιστεί ο τεμαχισμός της Alstom. Το 2014 πούλησαν τον κλάδο ενέργεια στην ε, General Electric, αμερικανική. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο να σωθούν οι θέσει εργασία, αλλά και η καινοτομία και η πόλη καινοτομία που εξαρτώνται από του χώρου παραγωγή. Γι' αυτό θα πρέπει το δημόσιο να βοηθήσει οπωσδήποτε τι ε, τις βιομηχανίες που ε, υπολειτουργούν ιδιαίτερα όταν είναι φάροι. Θα πρέπει ε, και οι υπουργοί βεβαίω να ασχολούνται με αυτά και όχι με τη σταδιοδρομία τους. Πού είναι ο τραπεζίτης Μακρόν, δεν τα είδα όλα αυτά. Ε, ανάμεσα σε δύο φωτογραφίσεις για έντυπα lifestyle δεν άκουγε ε, τις εκκλήσεις για βοήθεια των εργαζομένων. Και τους έδωσε και το λόγο του ο Μακρόν, μηδέν απολύσεις. Ορίστε, 2.000 κινδυνεύουν να απολυθούν 500 στο Μπελφόρ περίπου. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε στη βιομηχανία ένα κράτος με στρατηγικό σχεδιασμό, με μακροπρόθεσμους στόχου, αλλά και με το χέρι στην τσέπη για να τους πετυχάνει. Ευχαριστώ. Ο το λόγο. Το Φεβρουάριο του 2013 η αναδιάρθρωση της Κατερπιλάρ με 1.400 απολυμμένους και μέλλον για την επιχείρηση το οποίο διαφαίνεται. Όλοι οι εργαζόμενοι όμως αποφασίζουν να δεχθούν περισσότερη ευελιξία και το αποτέλεσμα είναι σήμερα να απολυθούν όλοι και να κλείσει το εργοστάσιο του Γκοσλή. Αδιαφορώντας για τους εργαζόμενους, αδιαφορώντας για τον κοινωνικό διάλογο και αδιαφορώντας για τις ε, πολιτικές ε, αρχές της χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, ούτε και η τελευταία που κλείνει μια επιχείρηση. Θα αναφερθώ εδώ σε αυτά που έλεγε ο Φιλίπ Μέστοκ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, που αναφερόταν στην Κατερπίλαρ σαν σε μια επιχείρηση που λειτουργεί με τις αρχές του βιοκαπιταλισμού. Βλέπουμε ότι λειτουργεί το σύστημα αυτό με υπεργολαβίες, με αναθέσεις σε εξωτερικούς φορείς και κάθε προσπάθεια αναδιάρθρωσης έχει αποτύχει. Πραγματικά η στήριξη με επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητο να γίνει σήμερα βάσει ενός βιομηχανικού σχεδίου και αυτό σε όλους τους τομείς, στην ενέργεια, στις μεταφορές αλλά και στον ψηφιακό τομέα. Πρέπει να στηρίξουμε τις βιομηχανίες μας. Βλέπουμε σήμερα την Κίνα να παράγει με πολύ χαμηλό κόστος και με μια ανταγωνιστικότητα την οποία εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει όλοι να παίξουμε με το ίδιους κανόνες του παιχνιδιού. Να σεβόμαστε το περιβάλλον όταν οι Κινέζοι δεν σέβονται τίποτα, κανένα πρότυπο και καμία προϋπόθεση περιβαλλοντολογική. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά να αξιολογήσουμε και το σύμφωνο σταθερότητας και να μπορέσουμε να φτάσουμε στα σωστά συμπεράσματα. Χρειαζόμαστε προσανατολισμούς και προοπτικές οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρεβόντα Λόν έχει το λόγο. Χαίρομαι, Πρόεδρε, που το κοινοβούλιο μας δείχνει σημάδια αντίδραση για αυτά τα κλεισίματα. Άλστον στον Περφόρ και κατέπλα στον Κεσλή. Δεν ειναι καλό συζήτηση, αλλά έχουμε να κάνουμε ένα διακυβόμενο ευρωπαϊκό, δηλαδή η υλοποίηση μια πραγματική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Πριν λίγου μήνε εδώ είχαμε θετήσει ένα ψήφισμα ζητώντα από την Κομισιόν να υποστηρίξει κυρίω και περισσότερο την συνδρομική μηχανία τη Ευρώπη μέσω κοντιλίων και σχεδίου Juncker. Πριν πέντε μήνες είχαμε ψηφίσει και το τέταρτο συνδρομικό πακέτο, το οποίο ενθαρρύνθηκε από τους κύκλους ομηχανίας μεταξύ αυτών και Αλστρομ, επειδή επέτρεπε μια εναρμόνιση κανόνων στην Ένωση. Η φωνή λοιπόν αυτή ακούστηκε και από το Κοινοβούλιο και από τι επιχειρήσει και από του πολίτε. Έχουμε να κάνουμε εδώ με την προστασία τη βιομηχανία μα, ενώπιον ενός ανταγωνισμού διεθνούς όλο πιο σκληρού. Έχουμε λοιπόν την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά επιχειρήσεων οι οποίε πρημοδοτούνται. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και την αποτυχία μιας δημοσιονομικής πολιτικής που φρενάρει τις επιχειρήσεις μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη ευελιξία αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη βιομηχανία μας. Αυτό είναι ένα βασικό διακύβευμα. Τέλος, αυτή η συζήτηση αφορά και την πρόσπιση των οικογένειων των αντρών και των γυναικών που πλήττονται. Αν οι κυβερνήσεις λοιπόν πρέπει να κάνουν κάτι, εξίσου πρέπει να κάνουν κάτι και οι βιομηχανοί, ώστε να προστατεύσουν αυτές, αυτά τα άτομα πέραν της ε, πολιτικής και της νοοτροπίας των κερδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Νίκολσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν δύο εβδομάδες είπε η ότι θα χαθούν 200 θέσει εργασία στην Βόρεια Ιρλανδία. Δυστυχώ αυτή η ανακοίνωση ήταν με μια σειρά ανακοινώσεων. Είχαμε την κατερπίλα, είχαμε τη Μισελέν με τεράστιε απώλειε. Το 2014 JTI 200 εργασία πάλι. Ξέρω ότι αυτές οι θέσεις εργασίας είναι εξειδικευμένων εργαζομένων. Θέσεις που ωφελούσαν τις τοπικές οικονομίες και, είχαν μεγάλες, και έχουν μεγάλες επιπτώσεις αυτές οι απώλειες στην τοπική οικονομία. Όπως ακούσαμε και από αλλού στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να εντοπίσουμε και να να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε για το μέλλον και θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε αυτούς τους διχασμούς που υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό ακριβώς εγώ και σαν αδελφοί μου και η επιχειρηματική κοινότητα ζητάμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες στην ε, Βόρεια Ιρλανδία για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Κύριε Νίκολσον, από τον κύριο Φωσολίκα υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουγα τον συνάδελφο Νίκολσον προηγουμένως για αυτό το θέμα. Να το ρωτήσω λοιπόν. Πώς γίνεται να κάνουμε επαναβιομηχανοποίηση όταν έχουμε να κάνουμε τόσες ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που προσφέρουν τόσα πολλά πλεονεκτήματα σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης και είναι ευθυνότερο να παράγει κανείς σε αυτές τις χώρες από το να παράξει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω το συνάδελφο για το ερώτημά του. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Από την Κομισιόν προετοιμάζουν μια αντίδραση σε σχέση και με αυτές τις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που ανέφερα. Τώρα δεν ξέρω και στη Γεωργία, ας πούμε, πόσες συμφωνίες μπορούμε να κάνουμε χωρίς ακριβώς να καταστρέψουμε αυτά που παράγουμε στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται όχι μόνο με τη ΣΕΤΑ και τη TTIP, αλλά και άλλε συμφωνίε με Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ συμφωνίε εμπορικέ που πρέπει να μα απασχολήσουν. Θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώ τι επιπτώσει θα έχουν και πώ η Ευρώπη θα μπορούσε ακριβώ να απορροφήσει όλε αυτέ τι επιπτώσει αυτών των συμφωνιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεσάρνες για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ Εύχομαι να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να μπορέσει και η Άλστον και η Κατερπίρα να παραμείνουν και να έχουν παραγγελίες και παραγωγή. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και για τις δύο αυτές επιχειρήσεις ε, οι ευθύνες είναι κατανεμημένες μεταξύ των επιχειρήσεων και των ε, αρχών. Τουλάχιστον για την Αλστόμ αυτό ισχύει επί χρόνια, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει επενδυτικό σχέδιο και σαφώς υπάρχει και εθνική ευθύνη. Υπάρχει όμως και ευρωπαϊκή ευθύνη, καθότι απουσιάζουμε εδώ και πολλά χρόνια από κάθε είδους καθοδήγηση και σχέδιο σε οικονομικό και βιομηχανικό επίπεδο. Πρέπει να δείξουμε ότι επιτέλους η Ευρώπη έχει αποφασίσει να υιοθετήσει ένα οικονομικό και βιομηχανικό σχέδιο. Πρέπει να δράσουμε και να μην είμαστε θύματα αποφάσεων άλλων. Πολύ καλό θα ήταν να συναντηθούν οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων στην Μπελφόρ, στην περιοχή αυτή, έτσι ώστε να στείλουν ένα μήνυμα ότι σκοπός της Ευρώπης είναι να βρεθούν θέσεις απασχόλησης και να υπάρξει πλήρης απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξαναδεί τους κανόνες του ανταγωνισμού. Σήμερα υπάρχει παγκόσμιος ανταγωνισμός και μας χρειάζονται μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε όμως να χρησιμοποιούμε τεχνικές και πολιτικές του παρελθόντος. Χρειαζόμαστε επίσης και ένα επενδυτικό σχέδιο δεκαπλάσιο από αυτό που έχουμε σήμερα, που θα βασίζεται στην καινοτομία και στην έρευνα και όχι σε ένα ε, ταμείο το οποίο δεν θα στοχεύει την βιομηχανική δραστηριότητα. Κοιτάξτε τι κάνουν οι Αμερικανοί το Κογκρέσο στην Αμερική προστατεύει τα συμφέροντα των Αμερικανών. Περιμένω να κάνουμε το ίδιο και στην Ευρώπη και να μην δίνουμε στην Κίνα το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς όπως κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Λεγιαρίκ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αρχίσουμε να συζητάμε από τη σοσιαλισ... Ε, την κοινωνική τη μετώπιση της παγκοσμιοποίησης. Όχι. Είναι ακριβώς το αντίθετο από την ευρωπαϊκή πολιτική εκβιομηχάνησης. Θα πρέπει να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις. Παράδειγμα, πώς μπορούμε να δεχόμαστε η Caterpillar αυτή τη στιγμή να απολύει ενώ θα πάρουν 1,4 δις η μετοχή της μέρισμα. Η Alstom γιατί δεν έχει μέλλον, ενώ ε, θα πρέπει να αναπτυχθούν οι επιβατικές και μεταφορές εμπορευμάτων με τα αυριανά τρένα. Τα τρένα του αύριο με τις νέες προδιαγραφές για το περιβάλλον. Υπόθηκε ότι έκανε η τράπεζα 80 ε, δις το μήνα, ποσοτική χαλάρωση το σχέδιο Juncker. Α χρησιμοποιηθούν για τι αυριανέ επενδύσει για τι εταιρείε αυτέ, α διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τι παραγωγικέ επενδύσει, για την εργασία, για την κατάρτιση στην Κατερπιλάρ, με συνεργασία εντός της Ευρώπης ε, ε, των ε, συνδρομικών επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται μια την άλλη. Δεν μπορούμε να βρούμε το αντίστοιχο του Airbus στο σιδηρόδρομο για το τρένο. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε τι θέσει όπω κάνουν άλλοι, βλέπε οι ΗΠΑ να δώσουμε το λόγο αλλά και την ισχύ ε, και ε, την εξουσία στους εργαζομένους για να διαχειρίζονται ήδη την επιχείρησή τους. Ευχαριστώ κύριο Ζηγενή Ξαντώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, απίστευτα πράγματα αυτά που συζητάμε κάθε τρεις και λίγο εδώ ε, τα βιομηχανικά. Κάθε φορά την ίδια διαπίστωση κάνουμε. Η λιτότητα έχει σταματήσει κάθε δημόσια επένδυση και παραγγελίες για να εργασία στα κράτη, υποδομές που είναι απαραίτητες και για την κοινωνία και για την οικονομία. Κάθε φορά τα ίδια συζητάμε για την έλλειψη μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής που τόσο ε, ικτρά μας λείπει. Και χρειαζόμαστε πραγματικά μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, γιατί μπορεί να υπάρχουν εθνικές πολιτικές που χωλένουν πάρα πολύ. Η Alstom σήμερα ε, ε, είναι ε, ένα πάρτι υποκριτών. Επίτηδες δημιουργούν αυτό το σκάνδαλο οι ηγέτες, οι θύνοντε τη επιχείρηση για να επέμβει το κράτος και το κράτος κάνει ό,τι το ανακαλύπτει. Το 2007 όταν κάναμε τη μεγάλη συζήτηση και διάσκεψη στο Γκρενέλ για το περιβάλλον θελήσαμε να προωθήσουμε τις ιδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Η κυρία Ροαγιάλ, υπουργό ε, Περιβάλλοντος, και οικολογίας ε, σκότωσε τον οικολογικό φόρο που είχε δισεκατομμύρια έσοδα ε, κάθε χρόνο για να χρηματοδοτεί το τραμ. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Μία ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική χρειαζόμαστε, ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο με τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τραμ και εμπορευματικέ μεταφορέ με το τρένο, που είναι και αποδοτικέ και συμφέρουσε και οικολογικέ. Και είναι απαράδεκτο αυτό παρά να ρίχνουμε την ευθύνη στα κράτη. Θα πρέπει να φύγουμε από τον αυτοκινητόδρομο και να περάσουμε από το σιδηρο... στο σιδηρόδρομο. Και οι πόλει μα που είναι αφόρητο πια να αναπνεύσει κανεί θα πρέπει να αναζωογονηθούν από το τραμ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μονό. Euh, Κυρία Επίτροπε, κύριε Ζαντό, θέλετε λιτότητα αλλά και ευρώ. Αντιφατικό αυτό. Η περιπτώσει Alstom και Caterpillar ακριβώ δείχνουν τι επιπτώσει του υπερνεοφιλελεύθερου μοντέλου στην Ευρώπη και τι κοινωνικέ επιπτώσει του. Αυτέ οι επίλεκτε βιομηχανίε επιβαρύνουν την βιομηχανοποίηση τη Γαλλία εδώ 25 χρόνια. Είχαμε την General Electric και ή είχαν υποσχεθεί θαύματα και πράγματα, τα οποία όμω δεν είδαμε και κοιτάξτε που φτάσαμε σήμερα. Είχαμε επιδοτήσει για τον ανταγωνισμό, είχαμε στρατηγικέ επιχειρήσει, οι οποίε όμω ε, υπολείπονται άλλων επιχειρήσεων εκτό Ευρώπη. Έχετε διαπράξει οικονομικά εγκλήματα ει βάρος των πολιτών. Η μόνη σα ε, ε, η λογική παγκοσμιοποίηση είναι ει βάρο των εθνών. Μόνο ένα μοντέλο εθνικού πατριωτισμού, πατριωτισμού με μια μακρόπνοη στρατηγική όπως προτείνει το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία, είναι η μόνη λύση για τη Γαλλία. Thank you. Next speaker is... Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντερ, επόμενος ομιλητής, δύο λεπτά. la κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είναι σημαντικό για μένα να αναφερθώ στην, στην περίπτωση της Άλστομ στο, στο Μπελφόρ, στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια έχει περίπου 500 τη εργασία. Είχαμε μια σύμβαση 30 τραμ. Η Γαλλία δείχνει έλλειψη οράματος και θετεί υποσχέσεις. Όμως όλα αυτά δεν θα πρέπει να μας κάνουν να παραβλέπουμε κάποια πράγματα και δεν θα πρέπει να μας τρέφει τον ένα εναντίον του άλλου. Οι δυσκολίε που αντιμετωπίζει η Alstom νομίζω είναι συμπτωματικέ μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική κάτω των προσδοκιών τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με το 20% του ΑΕΠ. Το Ευρωκοινοβούλιο πέρσι, μάλλον τον περασμένο Ιούνι, ψήφισε ένα ψήφισμα για την ανταγωνιστικότητα του σιδηρόδρομου. Κυρία Επίτροπε, η Κομισιόν θα ξεκινήσει ένα δομημένο διάλογο με τον κλάδο αυτό, επειδή η βιομηχανία του σιδηροδρόμου περιλαμβάνει 80.000 θέσει εργασία πανευρωπαϊκά. Δυστυχώ, οι επιχειρήσει μα πολύ συχνά πρέπει να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό υπερπροστατευμένο με ισχυρέ επιδοτήσει και με εργασία σε χώρε που επιβάλλουν δεσμευτικού δεσμευτικούς κανόνες μετατόπισης μηχανικής. Υπάρχει λοιπόν πρόσβαση στι αγορέ μα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό λοιπόν στι διαπραγματεύσει με την Κίνα, την Ιαπωνία και τι ΗΠΑ. Θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αφελεί και να προστατεύσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή αγορά με ένα εργαλείο αμοιβαιότητα για την αγορά μα. Εμεί θα σα υποστηρίξουμε σε αυτό. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε το σιδηρόδρομο να βυθιστεί όπω και άλλε βιομηχανίε, κυρία Επίτροπε. Θα πρέπει επιτέλου να υιοθετήσουμε μια φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαγιά είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το πλήσιμο της κατεπίλνες του Γκουσλή είναι 6.000 θέσεις απασχόλησης που θυσιάζονται για να ικανοποιήσουμε τα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Αμερική. Πολλές ε, ευρωπαϊκές ε, περιοχές πλήττονται από τέτοιες αποφάσεις. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, καθώς και να χαιρετήσω την αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θα πρέπει πραγματικά να επιβάλλουμε κυρώσεις αποφασιστικές σε όλους αυτούς οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις ε, να κλείνουν εργοστάσια, να αφήνουν άνεργους εργαζόμενους ενώ έχουν κέρδη. Η βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης θα πρέπει να βασίζεται στην έρευνα και στην καινοτομία. Θα πρέπει να σταματήσουμε τα μέτρα λιτότητας και να επενδύσουμε στην πραγματική οικονομία, να δημιουργήσουμε ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Τι περιμένουμε. Έχουμε σήμερα αντιμετωπίσει πολλά τέτοια ανθρώπινα δράματα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους στην Κατερπίλερ, καθώς και όλους αυτούς που εργάζονται μέσω των ε, εταιριών υπεργολαβίας. Και την ίδια ώρα να στηρίξουμε όλες τις μέχρι τώρα προσπάθειες ε, για κατάρτιση και στήριξη των εργαζομένων. Εδώ και δέκα χρόνια τα κέρδη της εταιρείας αυτής μεταφέρονται στην Ελβετία. Πριν πάρει την τελική απόφαση να αφήσει άνεργους τους εργαζόμενους που τόσα χρόνια εργαζόταν στα εργοστάσια της. Θα πρέπει πραγματικά να στηρίξουμε όλους αυτούς που βρίσκονται σήμερα σε αυτή τη θέση, αλλιώς θα έχουμε πάρα πολύ έντονες και βίαιες αντιδράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άντερσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως Ευρωβουλευτής υποστηρίζω ε, τους εργαζομένους ε, σε ένα εργοστάσιο που ε, στην εκλογική μου περιφέρεια απειλούνται με απολύσεις για τα ωφέλη των ε, μετόχων, ε, με μερίσματα. Για να σωθούν οι θέσει εργασία θα μπορούσαν να είχαν μεράσει τι θέσει σε διάφορε μονάδε παραγωγή, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρουν είναι οι εκατομμυρούχοι μέτοχοι που θέλουν το μέρισμά του. Ε, και ας καταστραφεί και ένα εργοστάσιο και ας απολυθούν εκατοντάδες ε, εργαζόμενοι και οικογένειες τους να βυθιστούν στην απόγνωση. Δυστυχώς ε, θέλουν ε, κυριαρχεί εδώ η απληστία και όχι η λογική. Δράματα έχουμε, αλλιώς αν δεν αλλάξει η κατάσταση δεν αλλάζει τίποτα στην εκλογική μου περιφέρεια γιατί ελέγχει η Βρετανική κυβέρνηση τον έλεγχο και δεν δέχεται τη χρήση του Ταμείου ε, Παγκοσμιοποίησης για τις απολύσεις εργαζομένων ε, στη Βόρεια Ιρλανδία. Ευχαριστώ πολύ στα Ιρλανδικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρίμοντ, παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. 6.000 είναι οι εργαζόμενοι, άνθρωποι, ε, πατεράδες, μητέρες, οικογενειών. Κλείνει η Κατερπιλάρ το εργοστάσιο στο Γοσλί και οι άνθρωποι αυτοί είναι στην ψάθα. Αυτό μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους, όχι βέβαια. Έγινε με δίκαιο τρόπο και σωστό, όχι. Και αγαπητοί μάνατζερ, αγαπητοί μέτοχοι Κατερπιλάρ, θα πρέπει να ντρέπεστε. Δεν έγινε με σωστό τρόπο. Γι' αυτό βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να βοηθήσουμε τους απολυμένους. Και αυτό πολύ συγκεκριμένα μπορεί να γίνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Μακροπρόθεσμα όμως, και αυτό έχει σημασία, θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικές συνθήκες πλαίσιο στην Ευρώπη για να διαφυλάσσονται θέσεις εργασίας και βιομηχανία. Τρία πράγματα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα. Πρώτον, καταπολέμηση ε, αυτής ε, της διαφυγής. Η Κατελπιλάρ πάει τα κέρδη στην Ελβετία, δεν φορολογούνται ε, και δεν επενδύουν στο Βέλγιο. Ε, στην Ευρώπη κανονικά εκεί που γίνεται η εργασία θα πρέπει να ε, καταβάλλεται και ο φόρος. Αυτή η αρχή είναι απλή, θα πρέπει μόνο να εφαρμόζεται. Και εμείς υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε αυτή την πρόταση. Δεύτερον, και μια ερώτηση. Είναι ευφυές δημόσιες επενδύσεις, για παράδειγμα σε βιομηχανικά πάρκα, να ε, γίνονται σχεδόν αδύνατοι με τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα. Όχι βέβαια, αυτό σκοτώνει την επένδυση. Έχω συγκεκριμένη ιδέα. Ας αλλάξουν οι λεγόμενες προδιαγραφές ΣΕΚ έτσι ώστε κράτη, περιφέρειες, δήμοι και κοινότητες να κάνουν ε, επενδύσεις που να μην πρέπει να ε, ε, τις αποσβαίνουν μέσα στον πρώτο χρόνο. Επίσης, τι θα κάνουμε για να παραμείνει η βιομηχανία στην Ευρώπη, δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα. Αυτό γίνεται με επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Εμείς χρειαζόμαστε στην Ευρώπη πολλές Silicon Valley, όχι μία. Μόνο έτσι μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις χώρες φθηνού ε, εργατικού κόστους. Θα πρέπει να είναι η αριστεία ε, και τα κλάστερ μεταξύ των πανεπιστημίων, ε, πράγμα που κάνει και το Πανεπιστήμιο στο Άχεν και με το διτό λεγόμενο σύστημα ε, εκπαίδευσης στην επιχείρηση και στο σχολείο. Αυτό το οφείλουμε λοιπόν στους εργαζομένους, στους απολυμμένους στον Κοσλή που ε, περιμένουν από εμά να τους βοηθήσουμε. Λόγια φτάνουν, έργα χρειάζονται τώρα. Η κυρία Βέρνερ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ε, να σας πω στοιχεία. 79-69 και πάνω από 30 χρόνια φτιάχνουν ε, μηχανές τρένων ε, στο Μπελφόρ και μηχανήματα κατερπιλάρ στην Κοσλή. Αν κλείσουν αυτά τα δύο εργοστάσια χάνουμε και know-how, τεχνογνωσία και ευρωπαϊκή βιομηχανική ιστορία. Για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους είναι πραγματική καταστροφή οι αποφάσεις των επιχειρήσεων. Κάτι όμως που ξεχνάμε συνέχεια στη συζήτηση είναι ότι δεν είναι μεμονωμένα αυτά. Έχει γίνει τάση από το 2008 μέχρι το 2014 3,5 εκατομμύρια έχουν χαθεί στη βιομηχανία. Μόνο στη Γαλλία από το 2000 έχει χάσει πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στη βιομηχανία ανταγωνισμός επιθετικός και κατά τα άλλα με κρατικές ενισχύσεις από Κινέζους και άλλους εκθέτει σε μεγάλη πίεση το σιδηρόδρομο και άλλους τέτοιους κλάδους. Υπάρχει και ψηφιοποίηση, ρομποτοποίηση ε, της ε, παραγωγής που μπορεί να είναι ευκαιρία για κάποιους αλλά απειλεί και θέσεις εργασίας. Και πού είναι η παραγωγικότητα. Ε, τρέχει πίσω από τις εξέλιξεις και την αγορά βιομηχανία ε, πιέζει τους εργαζομένους, τους αρρωσταίνει από την πίεση και χάνουμε και τη βιομηχανική μας βάση συνέχεια στην Ευρώπη. Τι σχέση έχει αυτό με κοινωνική οικονομία της αγοράς αξιόπιστη, τίποτα πια. Η γαλλική κυβέρνηση στην υπόθεση Αλστόμε επενεύει και καλά έκανε, αλλά το Παρίσι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο βασικό πρόβλημα δεν, δεν μπορεί να σωθεί μόνη της καμιά χώρα για να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Χρειαζόμαστε ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κοινά συμφέροντα να προωθούμε στην βιομηχανική μας πολιτική. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική χρειάζεται να διατυπώσουμε και να την ενισχύσουμε με κρατικά μέσα. Έχω αυτή την προσδοκία από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βιομηχανική πολιτική της ήρεμης δύναμης τώρα πια δεν πρέπει να έχει τελειώσει. Φτάνει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλήν. Ο Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί Επίτροπε, οι αρνητικές επιπτώσει των αποφάσεων για Άλστον και Caterpillar θα ακουστούν και στην Ιταλία, τη χώρα μου. Φαίνεται ότι ε, λόγω θέσης εργασίας της Άλστον στον Μιλάνο είναι πάνω από 200. Εύχομαι λοιπόν και η Ιταλική κυβέρνηση να συμμετάσχει στην προσπάθεια ανέβρεση λύση, γιατί ο αριθμός θέσεων εργασία είναι τεράστιος και για τη χώρα μου. Εξάλλου έχουμε και το θέμα της Ευθύνη της Ένωσης γενικότερα όσον αφορά τη δυνατότητα ανάκαμψη του μεταποιητικού τομέα. Το έχουμε ξαναπεί ότι η βιομηχανία και η μεταποιητική βιομηχανία δεν πρέπει να δέχεται παρεμβάσει ευρωπαϊκέ. Όμω πολλέ από αυτές τις παρεμβάσεις έχουν έμεσε επιπτώσει όσον αφορά την ανάκαμψη τη βιομηχανία. Να μην παραπονιόμαστε λοιπόν για την απώλεια θέσεων εργασία και μετά να κάνουμε πολιτικέ α πούμε στον τομέα τη ενέργεια που είναι τελείω αντίθετε με την ανάπτυξη τη βιομηχανία μα. Να μην παραπονιόμαστε για την απώλεια θέσεων εργασία και μετά να κλείνουμε το μάτι στην ε, Κίνα με την αναγνώριση της οικονομίας αγοράς και να μην παραπονιόμαστε για απώλεια θέσεων εργασία και μετά να κάνουμε παραχωρήσεις στους δημόσιους ε, προπολογισμού στις χώρες μας με στοιχεία τελείως αντίθετα που βαραίνουν δηλαδή την ανάκαμψη τη βιομηχανική των χωρών μας. Πρέπει λοιπόν σε συνεργασία κράτος και ιδιώτες να αποτελέσουν το γόνιμο έδαφος για την ανάκαμψη των οικονομιών μας και όλων των θέσεων εργασία που σχετίζονται με τις οικονομίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Λόπες. Πρέπει να επαναβιομηχανοποιήσουμε την Ευρώπη ώστε να έρχει ισχυρή βιομηχανία, γιατί αυτό σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη. Γιατί και βιομηχανία πρέπει να συνδέεται με καλές αμοιβέ, κοινωνική προστασία και σταθερές θέσεις εργασία. Για να επανοβιομηχανοποιήσουμε όμως την Ευρώπη, καταρχάς θα πρέπει να προστατεύσουμε τη μηχανία που ήδη έχουμε σήμερα. Εγώ έχω βαρεθεί στην Καταλωνία, στην ε, εκλογική περιφέρεια, να συναντώ όλους τους φορείς που υποφέρουν από μετασχηματισμούς, από κλεισίματα, από συγχωνεύσεις, όπως στην περίπτωση της Alstom, που και εκεί έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει δεχτεί αναθεώρηση εργασιακή πολύ επιθετική. Ξέρω ότι η Επίτροπο Τάισεν συμμερίζεται αυτές τις ευαισθησίες. Πρέπει όμως να δράσουμε. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε κοινού κανόνες που θα διασφαλίζουν και εξασφαλίζουν τους εργαζόμενους ενώπιον διαδικασιών όπως αυτές. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κοινοί κανόνες όσον αφορά τις διαβουλεύσεις που ισχύουν για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάτσε τώρα. Κέλλη, πρώτος ομιλητής. Να νομίζω είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση γιατί μία από τις προκλήσεις μας για να κάνουμε και πάλι την Ευρώπη ανταγωνιστική είναι η επαναβιομηχανοποίηση πέρα από το 2020. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Σταγέννη είχε πει ότι θα έχουμε μια βιομηχανία που θα είναι γεμάτη από μετεγκαταστάσεις με απώλεια θέσεων και εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλες δάσεις, όπως η μείωση και όχι η αύξηση του διεξιδίου των ρήπων και διεξιδίου του άθρακα. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για το μέλλον. Πάνω απ' όλα θα πρέπει να επαναβιομηχανοποιήσουμε την Ευρώπη και να βρούμε τον τρόπο για το κάνουμε αυτό. Σε σχέση και με τη συμφωνία του Παρισιού, είναι τεράστια ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας. Αν λοιπόν εμείς εφαρμόσουμε στόχους για να νεώσουμε ενέργεια και άλλους, έτσι θα συμβάλλουμε στις απαραίτητες μηχανικές επιτυχίες που χρειάζεται εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπλάνκο Λόπες, επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, το πρωί λέγαμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι κρίσεις αλυσοδένουν την Ευρώπη και αυξάνεται η δυσφορία των πολιτών Έχουμε αύξηση των ισοτήτων, έχουμε απώλεια εισοδημάτων και μισθών, απώλεια θέσεων εργασία, απώλεια απασχόληση. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ανάκαμψη τη βιομηχανική πολιτική στο σύνολο τη Ένωση. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα τηρήσουμε τον στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση τη βιομηχανία στο ΑΕΠ από το 15% στο 20%. Θα πρέπει να περάσουμε λοιπόν από τα λόγια στα έργα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και οπωσδήποτε βέβαια θα πρέπει να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping και τον αθέμητο ανταγωνισμό που έχουμε και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των χωρών μελών όπως στον τομέα του Χάλιβα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για την αντιστάθμιση των μηχανιών υψηλή κατανάλωση ενέργειας ώστε να μην μπορεί κάθε χώρα να κάνει τέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητή Επίτροπε, νομίζω ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να παραβλέψει την ανάγκη επαναβιομηχανοποίησης, η οποία αποτελεί μια ευκαιρία ενίσχυσης της εργασίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών μας. Γι' αυτό σας προτείνω να επιμείνουμε για τις πολιτικές άμυνας, τις εμπορικές, και αντιμετώπιση του αθέμη του ανταγωνισμού, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πιο περίπλοκη νομοθεσία και σκέφτομαι με τρόμο την διαφορά, ας πούμε, στι προδιαγραφέ παραγωγή των προϊόντων. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι για του κανονισμού. Θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να υπάρχει εθελούσια συμμόρφωση. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τη βιομηχανία. Υπάρχει άλλο ένα ζήτημα, το οποίο ανέκαθεν επεσήμανα στη δραστηριότητά μου μια πολιτική προάσπισης εμπορικής των ευρωπαϊκών προϊόντων αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά στην κλωστή φαντοργία, στην αυτοκινητοβιομηχανία ή στον χάλιβα. Αν θέλουμε λοιπόν την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης θα πρέπει να θέσουμε τέλος στον αθέμητο ανταγωνισμό σε αυτούς τους τομείς και στο τάμπινγκ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Πρόεδρε, η βιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα κυρίως μετά την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση. Τα τελευταία χρόνια στην Ένωση έχουν κλείσει εκατοντάδες μονάδες παραγωγής και έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας τώρα ήρθαν να προσθεθούν στη λίστα οι μονάδε και οι εργαζόμενοι τη caterpillar και τη alstom. να σημειώσουμε ότι και στην ελλάδα λόγω του μνημονίου και τη Τρόικα έκλεισαν χιλιάδε επιχειρήσει με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν στρατιέ ανέργων. πρέπει να αναγνωρίσουμε επίση ότι η caterpillar έκλεισε παρά το γεγονό ότι η εταιρεία είχε τηρήσει το στόχο συρρήκνωση κατά 36% του κόστου παραγωγή τη το δε εργοστάσιο της alstom έκλεισε μετά από την υπογραφή μεγάλου συμβολέου προμήθειας των γαλλικών σιδηροδρόμων από γερμανική εταιρεία. αυτά είναι τα αποτελέσματα της γερμανικής ευρώπης μιας ευρώπης της λιτότητας που μέχρι σήμερα δυστυχώς υπηρέτησαν με ευλάβεια η βελγική και γαλλική κυβέρνηση. επανεκβιομηχάνηση της ευρώπης δεν γίνεται όμως με συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου τύπου ttip με λιτότητα και με μια οικονομία υποταγμένη στις προσταγές του βερολίνου. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιάκοβτσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στο βιομηχανικό μας μοντέλο και το σχέδιο εκβιομηχάνησης της Ευρώπης. Τι είδους βιομηχανία θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι λίγα υπόθηκαν και λίγα άκουσα σήμερα όσον αφορά αυτό το μοντέλο. Θα πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όταν μιλάμε για την Alstom και για την Caterpillar. Βεβαίως και θα πρέπει να αντιδράσουμε και να δείξουμε αλληλεγγύη προς όλους αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους. Κάτι άλλο όμως που μας απασχολεί εδώ είναι τι θα γίνουν αύριο οι άνθρωποι αυτοί. Τι μοντέλο έχουμε να τους προσφέρουμε. Παραδείγματος χάρη ο κατασκευαστικός τομέας, τα ναυπηγεία, τα οποία πραγματικά είναι ευρωπαϊκό σχέδιο. Να μην καταστρέψουμε τα εναπομείναντα στον τομέα αυτό, στα ναυπηγεία και στην κατασκευή πλοίων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο, κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Σημείωσα τα περισσότερα από αυτά που μου προτείνετε. Η πρώτη μας προτεραιότητα, η άμεση προτεραιότητά μας είναι βεβαίως να συνοδεύσουμε και να στηρίξουμε αυτούς που πλήττονται άμεσα, να δείξουμε αλληλεγγύη με τους εργαζόμενους και τις περιοχές που πλήττονται από τα κλεισίματα αυτά και βεβαίως να στηρίξουμε με τα ταμεία και τα σχετικά εργαλεία που διαθέτουμε. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε μία πρόταση για να συνεχιστεί η επέκταση που προβλέπεται όσον αφορά την εξαίρεση άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στο σχέδιό μας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης να απλοποιήσουμε τους κανονισμούς και τις ρυθμίσεις με φορολογικά κίνητρα τα οποία να δίνουν έναυσμα, να δίνουν κίνητρα και να μην απογοητεύουν και δυσκολεύουν τις επενδύσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε και με άλλους τρόπους ε, θέσεις απασχόλησης εμβαθύνοντας ε, την ενιαία αγορά. Και η Ευρώπη γνωρίζουμε όλους ότι έχει τις δυνατότητες ε, να βελτιώσει την κατάσταση του τομέα της απασχόλησης και στον τρίτο πυλώνα του σχεδίου επενδύσεων να δώσουμε κίνητρα για καλύτερη και βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το κλείσιμο του εργοστασίου της Κατερπίλαρ στο Βέλγιο δεν αφορά άμεσα το σύμφωνο σταθερότητας. Είναι καθοριστικό αυτό το σύμφωνο για να στηρίξουμε και να δώσουμε κίνητρα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν εμποδίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης περαιτέρω επενδύσεις στην Ευρώπη. Όπως είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιούγκερ. Πρόκειται για ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, να στηρίξουν την ανάπτυξη. Και γνωρίζουμε το ψήφισμα στο οποίο αναφερθήκατε, προετοιμάζουμε μία απάντηση και φυσικά και σημειώνουμε όλες τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχονται σε αυτό το ψήφισμα. Σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε και να στηρίξουμε την βιομηχανία στην Ευρώπη. Μπορώ επίσης να σας πω ότι οι Επίτροπες Μάλστρομ είναι εν μέσω μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης. Είναι καλή διαπραγματεύτρια και σκοπός της είναι και παραμένει να στηρίξει αυτές τις επενδύσεις και να λάβει υπόψη της όλες τις κοινωνικές συνέπειες, να προσφέρει προοπτικές και ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Αναφερθήκατε και στην Κίνα και τον ανταγωνισμό. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική απόφαση για το θέμα αυτό. Αυτό που όμως σίγουρα ξέρω είναι ότι θα δημιουργήσουμε αποτελεσματικά εργαλεία για τις εμπορικές μας σχέσεις, κάτι το οποίο θα ενισχύσει και δεν θα αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα συνεχίσω στα γαλλικά, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μπαγιέ ότι και εγώ χαιρετίζω την αντίδραση των ε, συνδικαλιστικών ε, οργανώσεων που με πολύ αξιοπρεπή τρόπο αποφάσισαν να στηρίξουν τις προσπάθειες των εργαζομένων. Θα τους στηρίξουμε και εμείς. Η απόφαση της ε, διεύθυνσης της επιχείρησης είναι για μας ακατανόητη αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι γιατί πέρσι μόνο 9.300 θέσεις απασχόλησης σώθηκαν στην περιοχή της Βαλονίας. Πρόκειται λοιπόν εδώ για ένα εργοστάσιο σύγχρονο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Σαρλερουά, στην πρωτεύουσα του Βελγίου, στις Βρυξέλλες, και τα άτομα που πλήττονται από την απόφαση της Κατερπίλαρ μπορεί να μην τους αρκεί αυτή η είδηση αλλά είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε για να βρεθούν λύσεις για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Επίτροπε. Ε, κλείνει η συζήτηση αυτή. ψηφοφορία